και ούτε μπλε Και τώρα λοιπόν το λόγο να δώσω τώρα πρώτα η κυρία Λαϊμτότα Στραουγιούμα, Πρωθυπουργός της Λετωνίας. Παρακαλώ κυρία Στραουγιούμα. Αξιότιμα πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, αξιότιμη επίτροπε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Σούλτς για τη θαυμάσια συνεργασία που έλαβε χώρα. Είναι τιμή το ότι παρευρίσκομαι εδώ και πάλι μετά από έξι μήνες πολύ έντονης εργασίας για να συζητήσουμε τα επιτεύγματα της Λετωνικής Προεδρίας. Η περίοδος ήταν, είχε ιδιαίτερες προκλήσεις, ήταν δυναμική η περίοδος, ήταν περίοδος μεγάλης ευθύνης και ήταν μια μοναδική εμπειρία για τη Λετωνία. Η Λετωνία είχε θέσει τρει προτεραιότητες. Ε, ανταγωνιστικότητα για την Ευρώπη, ψηφιακή Ευρώπη και μια Ευρώπη που να συμμετέχει στου καθημερινού αγώνε. Η ζωή, ωστόσο, διόρθωσε τις αρχικές μας προβλέψεις. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις και η ανθρωπιστική κρίση στους, ε, στα σύνορα της Ευρώπης ε, χρειάζονταν άμεση ανταπόκριση από πλευράς μας. Ενώ τώρα οι σκέψεις μας όλες είναι με την Ελλάδα. Ναι μεν η Λετωνία ήταν επικεφαλής της ε, Προεδρίας του Συμβουλίου σε περίοδο σοκ και αβεβαιοτήτων. Είμαι περήφανη διότι η χώρα μου με επιτυχία επετέλεσε τα καθήκοντά της την πρώτη φορά που προέδρευσε της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μετά από 10 χρόνια συμμετοχής. Επιτύχαμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες και θα ήθελα να σημειώσω ιδιαίτερα ότι ένα συνεχώς παρόν στοιχείο κατά την Προεδρία μας ήταν η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και ο κοινωνικός διάλογος. Αξιότιμη Ευρωβουλευτής κατά την προετοιμασία και την εξαγωγή της Προεδρίας είχαμε έντονο διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι μας κάναμε κάθε προσπάθεια για να επιτύχει η Λετωνική Προεδρία και μόνο χάρη στη συνεργασία χέρι με χέρι όλων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μπορούμε να επιτύχουμε αποτελέσματα και να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ένωση. Από πλευράς της Λετωνικής Προεδρίας θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη θαυμάσια συνεργασία που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Αυτή η θαυμάσια και επικοδομητική συνεργασία μας βοήθησε να σημειώσουμε αποτελεσματική και ρεαλιστική πρόοδο σε όλα τα σημαντικά θέματα και μας επέτρεψε να αντιδράσουμε ταχαίως στις νέες προκλήσεις και κρίσεις που αντιμετωπίσαμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργαστήκαμε για μια σειρά νομοθετικών θεμάτων και σημειώθηκε πρόοδος ε, για διάφορα θέματα. Συμφωνήσαμε για σημαντικά θέματα και επιτύχαμε απτά αποτελέσματα. Τώρα, κάνοντας απολογισμό, θα ήθελα να τονίσω τις πιο σημαντικές επιτυχίες μας που ε, σημαίνουν ωφέλη για όλους τους πολίτες. Πρώτα απ' όλα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ΕΦΣΥ. Σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καταφέραμε να επιτευχθεί συμφωνία για το Ταμείο αυτό. Ήδη ε, τώρα το καλοκαίρι θα αρχίσει να λειτουργεί το Ταμείο και θα προσελκύσει επενδύσεις προς την Ευρωπαϊκή Οικονομία. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, ιδιαίτερα έντονη και σκληρή εργασία για το θέμα αυτό, που είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη. Δεύτερον, ενεργειακή ένωση. Θέσαμε τα θεμέλια για την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση για να ενισχύσουμε την ενεργειακή μας ανεξαρτησία και για μια κοινή ενεργειακή πολιτική. Κατά την εργασία μας εστιάσαμε στην αναγκαιότητα διασφάλισης σταθερής ε, ενέργεια σε λογικές, σε βατές τιμές για τους καταναλωτές για να υπάρξει καλύτερη πληροφόρηση για τους προμηθευτές ενέργειας για όλους. Η Λετωνική Προεδρία επέτυχε να ληφθούν ουσιώδεις αποφάσεις για να τεθούν λοιπόν τα θεμέλια της Ενεργειακής Ένωσης. Έτσι προθίσαμε επίσης την μετάβαση σε μια ενέργεια χαμηλού άνθρακα και αυτό σημαίνει ότι προωθούμε και το στόχο της ενεργειακής ανεξαρτησίας. Χαιρόμαστε που επετεύχθη συμφωνία για συγκεκριμένους στόχους για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μετά το 2020. Έτσι, συμβάλλουμε στην επιτυχία της διάσκεψης ε, των Παρισίων. Επίσης, ψηφιακή αγορά. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να συμβαδίζουμε με την πρόοδο της τεχνολογίας, ούτω ώστε η κοινωνία μας να μπορέσει να προσαρμοστεί στην ψηφιακή εποχή. Συμφωνήσαμε λοιπόν μια σειρά από μέτρα που θα προωθήσουν τη χρήση ψηφιακών λύσεων για τις επιχειρήσεις. Είναι θέματα και πρόσβασης και ασφάλειας δεδομένων και βεβαίως την προώθηση και απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Επίσης ασχοληθήκαμε με την πλήρη αξιοποίηση της ψηφιακής οικονομίας από την, ε, της ψηφιακής οικονομίας για την κοινωνία μας γιατί όλα αυτά θα είναι κρίσιμη σημασία για την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ένωση. Η Λετωνική Προεδρία έκανε ό,τι μπορούσε, ό,τι ήταν δυνατόν για να προωθηθούν ε, τα ευαίσθητα ε, νομικά κείμενα που θα προωθήσουν την ψηφιακή αγορά. Και χαίρομαι που το Συμβούλιο ενέκρινε τη γενική προσέγγιση για τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, κάτι που επιτρέπει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που όντω ξεκίνησαν στι 24 Ιουνίου. Είναι ουσιώδη προπόθεση αυτό για να αναπτύξουμε την ε, ενιαία ψηφιακή αγορά και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών μα. Τις τελευταίες ημέρες της Προεδρίας επετέφθη συμφωνία και για την πρόταση για την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών. Αυτό θα επιτρέψει την κατάργηση των τελών περιαγωγής και θα διασφαλίσει την ε, ανοιχτή πρόσβαση στο ίντερνετ. Αυτό είναι ουσιώδης επιτυχία της Προεδρίας μας και θα ωφελήσει όλους τους πολίτες, διότι αυτή η συμφωνία επιτρέπει ουσιώδη μείωση ήδη στα τέλη περιαγωγής, ήδη από τι 30 ε, Απριλίου του 2016 επίσης επετέφθη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τι ε, γενικέ αρχέ για την ασφάλεια του δικτύου και των πληροφοριών, την ε, οδηγία NIS. Και είμαι πεπισμένη ότι όταν θα καταλήξουμε στα τεχνικά θέματα θα έχουμε το πλαίσιο που θα επιτρέπει καλύτερη προστασία από τι επιθέσει των κυβερνοχώρο. Τέταρτον, μετανάστευση. Του τελευταίου μήνε η μετανάστευση έχει γίνει τα πιο σημαντικά και τα πιο επίκαιρα θέματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση η εφαρμογή της, ε, των οδηγιών των κατευθυντηρίων οδηγιών που έχει συμφωνήσει το Συμβούλιο ήταν αναγκαία για να καταπολεμήσουμε τους διακινητές, να μειώσουμε τους θανάτους του Μεσόγειο και να ε, συνεννοηθούμε με τις χώρες προέλευσης και μετάβασης ούτως ώστε να βοηθήσουμε τις χώρες που υφίσταται την περισσότερη μεταναστευτική πίεση. Είναι πολύ περίπλοκο το θέμα της μετανάστευσης. Και μια μόνιμη και βιώσιμη λύση μπορεί να γίνει μόνο εάν υπάρξει μια ολιστική και ισορροπημένη και επίμονη αντιμετώπιση, ούτως ώστε να έχουμε μια συστηματική και σταδιακή εφαρμογή. Όσον αποφασίζονται, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι λύσεις που θα επιδιώξουμε να εφαρμόσουμε στηρίζονται από όλα τα κράτη-μέλη. Πρέπει να βρούμε την, αλληλεγγύη, συγγνώμη, την ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύη και υπευθυνότητα. Και τα δύο είναι ουσιώδη τμήματα τη μεταναστευτική πολιτική τη Ένωση. Πρέπει να χορηγήσουμε προστασία σε όσους τη χρειάζονται. Ωστόσο, τα μέτρα προστασίας δεν θα αρκέσουν από μόνα τους. Πρέπει να συμβαδίζουν με ένα αποτελεσματικό σύστημα επιστροφής των παρατύπων μεταναστών. Πέμπτον, ασφάλεια. Οι προκλήσεις ε, στον τομέα αυτό μας έκαναν να επανεξετάσουμε την εσωτερική και εξωτερική μας ασφάλεια. Κατά την Προεδρία μας επετέχθησαν αρκετά για να ενισχύσουμε την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης. Τον Ιούνιο οι Υπουργοί Εσωτερικών ενέκριναν μια ε, ανανεωμένη στρατηγική εσωτερική ασφάλεια που θέτει προτεραιότητε για την προσεχή πενταετία, οι οποίε είναι κατά καταπολέμηση τρομοκρατία και τη ρίζο παστικοποίηση πολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο και των κύβερνων επιθέσεων, Όλα αυτά ε, καταδεικνύουν ποιε είναι οι νέε προκλήσει που αντιμετωπίζουν στην ασφάλεια. Για παράδειγμα, υβριδικέ απειλέ τι ε, τελευταίε εβδομάδε. Για άλλη μια φορά ε, ε, διαπιστώσαμε πόσο επίκαιρε είναι αυτέ οι απειλέ. Και ε, σα υπενθυμίζω ότι τηρήσαμε στο Συμβούλιο την υπόσχεσή μα να συμφωνήσουμε για το πακέτο για την προστασία των δεδομένων. Και πραγματικά ελπίζουμε ότι μέχρι τέλο του χρόνου θα είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε για το Μητρό ε, Στοιχείων των Επιβατών της Ένωσης, το PNR. Αναγνωρίζουμε ότι η συμμετοχή της ε, υπάτης εκπροσώπου στην αναθεώρηση της στρατηγικής ήταν επίσηματική. Έκτον, ανατολική εταιρική σχέση. Χαιρόμαθε ιδιαίτερα που η συνάντηση κορυφή στη Ρήγα προώθησε σταθερές σχέσεις ε, της Ένωσης με τους εταίρους της Ανατολικά Σημειώνουμε ωστόσο ότι υπάρχει μια διαφοροποιημένη προσέγγιση που θα είναι σημαντική στο μέλλον. Και θα είναι σημαντικό να κατοχυρωθεί η ανατολική εταιρική σχέση μαζί με το, με το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Προεδρία επέτυχε συμφωνία για μικρό χρηματοπιστωτική στήριξη στην Ουκρανία. Και χαιρόμεθα και χαιρετίζουμε το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε ενωμένη για το θέμα της Ρωσίας και συνέχισε να τονίζει πόσο σημαντικό είναι να ε, γίνουν σεβαστές οι συνθήκε του Μίνσκ. Κατά την Προεδρία μας, βασικό ρόλο έπαιξε και πάλι οι σχέσεις μας με την Κεντρική Ασία. Δεν πρέπει να υποτιμούμε την περιοχή αυτή. Έβδομον, TTIP. για την ανάπτυξη της οικονομίας μας είναι πολύ σημαντικό να προσελκύσουμε επενδύσεις και να προωθήσουμε επίσης και το εξωτερικό εμπόριο. Γι' αυτό είναι ουσιοδέστατο να καταλήξουν έγκαιρα οι διαπραγματεύσεις Ένωσης, είπα, για αυτήν την ολιστική και αμοιβαία εποφελή συμφωνία που είναι η Διατλαντική Συμφωνία για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις. Το TTIP θα το συζητήσετε φυσικά ως επόμενο θέμα στην μέση διαταξή σας. Και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας στηρίξει ε, στην προσπάθεια ολοκλήρωσης αυτών των διαπραγματεύσεων γιατί αυτή η συμφωνία δεν θα παίξει μόνο οικονομικό αλλά και ουσιοδέστατο γεωστρατηγικό ρόλο. Μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργαστήκαμε έντονα και για διάφορα άλλα θέματα που είναι πολύ σημαντικά για την ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για το ότι μας βοηθήσατε να εστιάσουμε σε αυτά τα θέματα και ορισμένα μάλιστα ορισμένες πλευρές ε, της πολιτικής απασχόλησης που είχαν περάσει το περιθώριο λόγω της οικονομικής κρίσης. Εστιάσαμε λοιπόν συγκεκριμένα στο ότι χρειάζεται ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ότι πρέπει να υπάρχουν βιώσιμες θέσεις εργασίας και δυνατότητες εξέλιξης στα διαδρομία των εργαζομένων. Και επιτύχαμε συμφωνία για να επιταχυνθεί η χρηματοδότηση των προγραμμάτων για την απασχόληση των νέων. Ένα δις ευρώ είναι διαθέσιμο για το πρόγραμμα αυτό, ούτως ώστε να βοηθήσουμε 650.000 νέους κάθε χρόνο. Θα ήθελα επίσης να μιλήσω για το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό πακέτο, τη συμβατότητα και την ασφάλεια. Και αυτό θα ωφελήσει <clears throat> όλους τους πολίτες και τον κλάδο. Και τον κλάδο. Οι καινοτομίες θα ε, προστατευτούν ε, λόγω της αναθεώρησης του συστήματος ε, διπλωμάτων έβρεση τεχνίας. Και θα λάβουμε και άλλα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών. Συμφωνήσαμε για διάφορα νομοθετήματα στον τομέα της γεωργίας, της προστασίας της υγείας και άλλων τομέων. Και χαίρομαι ότι στις 25 Ιουνίου τα τρία θεσμικά όργανα ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις για μια νέα διοργανική συμφωνία. Αυτό είναι μοναδική ευκαιρία για τα όργανα της Ένωσης να βελτιώσουν να τελειοποιήσουν τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Οι πολίτες μας αναμένουν αποτελεσματική λειτουργία από του θεσμού της Ένωση και είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι προσδοκίες θα γίνουν πραγματικότητα. Η Λετωνική Προεδρία έχει συνεργαστεί με έντονο και στόχο προσιλωμένο τρόπο για να επιτύχουμε μια ανταγωνιστική, ψηφιακή, ασφαλή Ευρώπη. Ε, εργαστήκαμε μαζί σου, Μάρτιν, και με τα άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνεργαστήκαμε στενά. Επίση με, με, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ζων Κλοντ. Και ελπίζω η ρεαλιστική μα προσέγγιση να έχει δημιουργήσει ένα σταθερό έδαφο για την επίλυση διαφόρων θεμάτων κατά τις επόμενες επιτυχείς προεδρίες. Και με αυτό το αίσθημα ότι τα πήγαμε καλά, περνάμε τώρα τη σκητάλη στην και Προεδρία. του. εύχομαι κάθε επιτυχία. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πιο δυναμικός και διασυνδεδεμένος. Και αυτό βεβαίω σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις αλλά και νέες ευκαιρίες προκύπτουν. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εργαστούμε με στοχοπροσιλωμένο τρόπο και αποφασιστικό και μόνο μέσω της συνεργασίας τα τρία όργανα μπορεί να επιτύχουν την επιτυχία των Ευρωπαϊκή Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο πρόεδρο κ. Γιούγκερ. Αξιότιμο κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα από καρδιάς να αποτίσω φόρο τιμή στο έργο το οποίο επιτέλεσε η Λεπτονική Προεδρία. Όπως είπατε και εσείς η ίδια κυρία Πρωθυπουργέ ήταν η πρώτη Προεδρία της Λετωνίας. Και για μια πρώτη Προεδρία πραγματικά τι εμπειρία, τι απόδοση. Σας ευχαριστούμε εξ ονόματος της Ευρώπης. όσοι δεν αγαπούν την Ευρώπη σίγουρα δεν μπορούν και να κάνουν κομπλιμέντα στους υπηρέτες της Ευρώπης, ε, σε όσους υπηρετούν την Ευρώπη. Κάνατε υποδειγματική δουλειά και θέλω να αποτίσω φόρο τιμή στις προσπάθειές σας και στα επιτεύγματά σας. Όλο ιδιαιτέρως θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, διότι πραγματικά ασχοληθήκατε με προσήλωση και αποφασιστικότητα με ορισμένα στήματα τα οποία είχαμε γύρει ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αμέσως μόλις αναλάβατε καθήκοντα και στη διάρκεια της, ε, του εξαμήνου σας, ιδίως ό,τι αφορά το σχέδιο επενδύσεων. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία ε, μεταξύ ε, των τριών θεσμικών οργάνων και καταφέραμε να φέρουμε σε αίσιο πέρας μέσα σε λίγους μήνες το φιλόδοξο αυτό σχέδιο. Ποτέ φόρο τιμή σε εσά, βέβαια, ποτέ φόρο τιμή ταυτόχρονα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το οποίο έδειξε και αυτό την αποφασιστικότητά του όποτε χρειάστηκε. Και επειδή μιλάμε για φιλοδοξίες, ούτε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίστασε να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις ορισμένες εξ των οποίων τι αναφέρατε, η ψηφιακή ένωση, η ενεργειακή ένωση, η ένωση των κεφαλαίων αγορών και ούτω καθεξής. Πλούσια, πλούσια και φιλόδοξη Προεδρία. Θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής όμως ε, και στο διαπραγματευτικό σας ταλέντο. Είναι γεγονός ότι από την έναρξη ισίω τη συνθήκη τη Λισαβόνα, ο ρόλο των Πρωθυπουργών και των Υπουργών Εξωτερικών έχει κάπω αλλάξει. Έχουμε τη μόνιμη Προεδρία του Συμβουλίου. Επομένω δεν προεδρεύει πλέον ακάστοτε ε, προεδρεύουν πρωθυπουργός. Ε, υπάρχει ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έχουμε τον ε, πρόεδρο ε, για, το για το Συμβούλιο Εξωτερικών και οι Υπουργοί Οικονομικών επίση έχουν δει το έργο του κάπω να ε, μειώνεται. Στην ε, περίπτωση του Λουξεμβούργου, εγώ έχω προεδρεύσει βέβαια και ε, το Eurogroup και το ECOFIN και αναλαμβάνουμε και τη Λουξεμβουριανή Προεδρία τώρα. Αυτή τη φορά είναι διαφορετικά τα πράγματα. Γνωρίζω πάντως ποια είναι τα υπέρ και τα κατά. Εσείς τα καταφέρατε με πολύ μεγάλη κομψότητα θα έλεγα ε, και πραγματικά θέλω να σας ε, συγχαρώ για το εξαιρετικό υποδεγματικό ε, έργο, κομψό έργο και εμείς μπορεί να είμαστε ευφυείς, αλλά υπάρχουν άνθρωποι πίσω από εμάς που κάνουν την πραγματική δουλειά και χωρίς αυτούς δεν είμαστε τίποτε. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Και θέλω και στη δημόσια διοίκηση, στους υπαλλήλους μας, να αποτίσω φόρο τιμής, γιατί και αυτοί κάνουν εξαιρετική δουλειά. Απόψε έχουμε ένα ακόμη Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ελλάδα, για το ελληνικό ζήτημα. Και να πω μερικά λόγια επίσημα γι' αυτό. Διαβάζω στο γερμανικό τύπο ότι ο Γιούγκερ ε, κρύβεται. Αλλά να μην χαίρεστε ήδη εκ των προτέρων πολύ. Για το ελληνικό δημοψήφισμα δεν είπα τίποτα ούτε την Κυριακή το βράδυ ούτε χθε. Γιατί ορισμένε φορέ πρέπει να γίνεται καμιά φορά αυτό. Πρέπει να σκεφτόμαστε πριν παίρνουμε τον λόγο. Και αυτό ισχύει και ορισμένου που φωνάζουν εδώ πέρα. Όχι, δεν κρύβομαι. Θα μιλήσω για πρώτη φορά για το ελληνικό ζήτημα εδώ, γιατί εδώ είναι ο χώρος της δημοκρατίας. Σε διάφορες ε, συνεντεύξεις μπορεί να μιλήσει κανείς, αλλά δεν αντικαθιστά αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ρόλο του. Εδώ θέλω να μιλήσω, γιατί τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει. Εδώ πρέπει να λογοδοτήσω, εδώ πρέπει να σας παρουσιάσω την άποψή μου. Λέγοντας το εξής. Δεν ήθελα να ξεκινήσω με αυτό, αλλά θα ξεκινήσω με αυτό. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πολλές φορές είναι αντικείμενο επικρίσεων για τα θέματα της Ελλάδας σε ορισμένα κράτη-μέλη. Ορισμένα μάλιστα γερμανικά μέσα ενημέρωση. Και ε, θα, ήθελε, θα ήθελαν ορισμένοι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι ένα πολιτικό όργανο και να εκφράζεται ε, πολιτικά. Ενώ άλλοι θέλουν να αποτελείται από ε, ουδέτερους υπαλλήλους ψηλού επίπεδου. Δεν είμαι ουδέτερος υψηλού επίπεδου ε, δημόσιο υπάλληλο. Είμαι πολιτικός. Και το βρίσκω καταπληκτικό, περίεργο, ότι για τα θέματα της Ελλάδας και του μέλλοντος της Ευρωζώνης όλοι μπορούν να μιλάνε κατά τη γνώμη ορισμένων και όχι ο πρώτος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα επιτρέψουν να με φημώσουν. Και το ίδιο ισχύει, θέλω να προσθέσω αμέσως, το ίδιο ισχύει και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τακτικά συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ε, μας παρουσιάζει τις απόψεις, τις ευαισθησίες, τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό το κάνει με πολύ ευχάριστο, αν και δεν είναι πάντα πολύ ευχάριστος για όλους, η αντίληψη ότι ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έρχεται στο Συμβούλιο παρουσιάζει κάτι, βγαίνει και μετά δεν θα πρέπει να ξαναμιλάει μέχρι να ξαναμπεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είναι πολύ περίεργη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι χάρτινος τίγρης. Και ασχολείται με τα θέματα της Ευρώπης και μεταξύ των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πολύ συχνά από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακόμη ε, και αν δεν έχει πάντα ε, σαφή εντολή, γιατί και εγώ δεν έχω πάντα σαφή εντολή για όλα τα θέματα, ορισμένε φορέ διευκρινίζει, ορισμένε φορέ με τρόπο έντονο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι χάρτινο τίγρη και ο πρόεδρό του δεν είναι λακέ κανενό. Μπορεί να μιλάει. Σήμερα το απόγευμα θα έχουμε άλλη μια συνάντηση κορυφής, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για την ε, υπόθεση της Ελλάδας. Καλό είναι αυτό όλοι λένε ότι πρέπει να σεβαστούμε την ψήφο του ευρωπαϊκού λαού. Και εγώ τη σέβομαι. Αλλά, αλλά, καταλαβαίνω την ψήφο τους. Γιατί ετέθη ένα ερώτημα ενώπιον του ελληνικού λαού που δεν μπορεί να τίθεται. Διότι τους πρότεινα να ψηφίσουν Κοιτάξτε, θα ήθελα να σας ρωτήσω εσάς, να μου πείτε αναλυτικά τι ερώτημα τέθηκε. Αλλά ας μην παρακάνουμε την ε, ε, διασκέδαση εδώ μέσα. Πρόεδρος. Περιμένετε παρακαλώ, λέει ο πρόεδρος κύριε. Περιμένετε παρακαλώ κύριε Γιούνκερ. Ο κύριος Γιούνκερ. Ε, νομίζω ότι τώρα ηρέμησαν ορισμένοι. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Παρακαλώ, λέει ο πρόεδρος, παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε ε, να ε, κάνετε κάποιες ε, παρατηρήσεις, αλλά δεν είναι δυνατόν να διακόπτετε τόσο πολύ τον ομιλητή. Κύριε Γιούνκερ, παρακαλώ, συνεχίστε. Δεν με, δεν με ευχαριστεί να με διακόπτουν ορισμένες φορές, με ευχαριστεί να με διακόπτουν αυτοί που πάντα διακόπτουν. Έλεγα λοιπόν πρέπει να συζητήσουμε πολύ συγκεκριμένα τι σημαίνει να σεβαστούμε την ψήφο των Ελλήνων. Και επειδή θεωρώ το θέμα σημαντικό, να πούμε σε τι είπαν όχι οι Έλληνες. Η πλειοψηφία των Ελλήνων είπε όχι για ένα κείμενο των τριών θεσμικών οργάνων, το οποίο είχε ήδη ξεπεραστεί κατά πολύ όταν τέθηκε σε ψηφοφορία. Μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη είχα έντονες διαπραγματεύσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και την ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ξέρει πολύ καλά ότι αυτό το οποίο υπευλήθη για ψήφιση στους Έλληνες δεν ήταν το κείμενο που ανταποκρινόταν στην κατάσταση των διαπραγματεύσεων. Και γι' αυτό σήμερα το απόγευμα, όπως και το προηγούμενο βράδυ, θα καλέσω τον Έλληνα Πρωθυπουργό να μου δώσει μια εξήγηση του τι σημαίνει αυτή η ψήφος. Γιατί το ερώτημα επί του οποίου χρειάστηκε να απαντήσουν οι Έλληνες είχε ξεπεραστεί κατά, πολύ και αυτό το ξέρουν όλοι όσοι συμμετείχαν σε διαπραγματεύσεις. Αλλά δεν είναι τόσο πολύ θέμα εδώ να μπούμε τώρα σε νομικίστικες λεπτομέρειες. Το μικρό μας εγώ και το μεγάλο δικό μου εγώ πρέπει να το βάλουμε σε δεύτερη μοίρα και να ασχοληθούμε με το θέμα που είναι ενώπιόν μας. Ποια είναι η κατάσταση. Όπως και πριν θεωρώ και θα συνεχίσω να το θεωρώ ε, μέχρι τέλους το αίτημά μου και η βούλησή μου είναι να αποφευχθεί ένα Brexit, να αποφευχεί, αποφευθεί έξοδο της Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Είμαι κατά ενός Brexit. Υπάρχουν κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ανοιχτά είτε και καλυμμένα είναι υπέρ μιας εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Έχω εμπειρίες από τη ζωή μου. Η εμπειρία είναι ότι οι απλές απαντήσεις είναι συνήθως οι λανθασμένες απαντήσεις. Είμαι κατά των απλών απαντήσεων. Για τα θέματα της Ευρώπης δεν υπάρχουν απλές απαντήσεις. Η Ευρώπη είναι η συνεχής προσπάθεια για συμβασμούς, για συμβαστικές λύσεις. Και αυτό είναι το καθήκον που έχει θέσει για τον εαυτό της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συνεχίσει να τον θέτει. Αυτό που θα ήθελα θα ήταν Ελλάδα. Αυτό το μεγάλο ελληνικό έθνος να μην έχει την εντύπωση ότι θέλουμε να βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς δεν μπορεί να θέλει να πετάξουμε την Ελλάδα έξω από την Ευρώπη. Και επειδή έτσι έχουν τα πράγματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει κάθε προσπάθεια ούτως ώστε οι διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα να επανεκκινήσουν. η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήμασταν εάν σταματάγαμε απότομα να συζητάμε. Εάν σταματήσουν τα ευρωπαϊκά ε, έθνη να συζητούν μεταξύ τους, τότε θα βαδίσουμε προς την ε, διάλυση της Ένωσης. Ήρθε νομίζω η ώρα, ούτως ώστε αυτή με κατανόηση και με λογική, αλλά και επίσης με ενθουσιασμό γιατί χωρίς συνέστημα δεν γίνεται τίποτα, θα πρέπει να προχωρήσουν. Λυπάμαι ιδιαίτερα που η ελληνική αντιπροσωπεία εγκατέλειψε την Τράπεζα των Ευρωπαϊκών. Δεν κάνει κανεί τέτοια πράγματα στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη διαπραγματεύεται κανεί μέχρι το τελευταίο χειριστό του δευτερολέπτου. Δεν το έκανε αυτό η ελληνική αντιπροσωπεία και αυτό είχε πολύ σοβαρέ επιπτώσει. Πρέπει και πάλι να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι. Αυτό πρέπει να είναι αυτονόητο για Ευρωπαίους και να επιχειρήσουμε να βρούμε μια λύση. Η λύση αυτή δεν θα προκύψει σήμερα. Γιατί αν προέκυπτε σήμερα θα ήταν μια υπεραπλουστευμένη λύση. Πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο για να γίνουν συζητήσεις και μέσω αλληλοκατανόησης και μέσω αποδοχής του ενός και του άλλου να διορθώσουμε την κατάσταση. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει επίσης θα πρέπει να σταματήσουν ε, οι ρητορικέ κορώνες. Να σταματήσουν απότομα μάλιστα να πω εδώ, εδώ στο ναό της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, δεν δέχομαι οι των θεσμικών οργάνων και δεν το αποδέχομαι και ως πρόεδρος της Επιτροπής να αποκαλούνται από την ελληνική κυβέρνηση τρομοκράτες. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται στην Ευρώπη. Όλοι προσπαθήσανε και κανένας δεν προσπάθησε όσο εμείς να αποφύγουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν θα τα ξαναπούμε και θα προσπαθήσουμε μέσω διαπραγματεύσεων χωρίς ρητορικέ ε, κορώνες να προωθήσουμε την κατάσταση και να καταλήξουμε σε μια συμφωνημένη λύση. Η Κομισιόν με κάθε σεβασμό για το αποτέλεσμα της ψήφου θέλει να μάθει τι σημαίνει αυτή η ψήφος. Δεν είναι όχι στην Ευρώπη, έτσι μου λέγεται, δεν είναι ναι προς το ευρώ, έτσι μου λένε. Άρα δεν μπορεί να είναι όχι και στις προτάσεις των θεσμών, γιατί δεν υπάρχουν αυτές τις προτάσεις. Πρέπει να τονίσουμε σαφώς ότι το μπαλάκι είναι στο γήπεδο της Ελλάδας. Πρέπει να μας εξηγήσουν ποιες είναι οι απόψεις τους σε αυτή την περίπλοκη κατάσταση. Πώς θα βγούμε από αυτήν. την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά της και ο Πρόεδρός της είναι διατεθειμένος να κάνει ό,τι είναι δυνατόν ούτω ώστε εντός αποδεκτών χρονικών ορίων να καταλήξουμε σε συμφωνία. Οι Έλληνες και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι μπορούν να βασιστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής για την ομάδα του έργου κύριος Βέμπα. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ την Προεδρία του Συμβουλίου για την επετελεστή συνεργασία, περιαγωγή προστασία των δεδομένων, ανατολική συνεργασία και πάνω απ' όλα το, η συμφωνία για τις επενδύσεις είναι θαυμάσιο αποτέλεσμα. Θαυμάσιος απολογισμός, σας συγχαίρω. Συγχαίρω ιδιαίτερα την κυρία Με Ευχαριστώ πάρα πολύ για το σταθερό χέρι, για τον ανθρώπινο τρόπο. Έχετε μια σύγχρονη κυβέρνηση στη Λετωνία, γιατί όπως βλέπετε στις πρώτες, στις πρώτες τρεις γραμμές κάθονται μόνο γυναίκες. Σας συγχαίρω για το πόσο σύγχρονη είναι η Προεδρία σας και εμείς Έχουμε και στο Προεδρείο του ΕΛΚ και μεταξύ των Ευρωβουλευτών 50% γυναίκε. Σα δάμε συγγνώμη γιατί λέμε πολλά για την Ελλάδα, αλλά θα έχετε σίγουρα κατανόηση γι' αυτό. Και μπορούμε να τα συνδέσουμε τα θέματα αυτά. Ότι η Λετωνία επίση πέρασε στο παρελθόν δύσκολε καταστάσει πριν από μερικά χρόνια. 14% μείωση του ΑΕΠ ε, ε, έχει το θάρρο η Λετωνία να κάνει και περικοπέ. Και σήμερα η Λετωνία έχει 2% ανάπτυξη συμβάλλει στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Επανήλθατε στην ορθή οδό. Και αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να πούμε. Μπορούμε να καταγγέλουμε την λιτότητα ή ό,τι θέλετε. Αλλά εάν δεν υπάρχει βούλη στην Ευρώπη για εσωτερικέ μεταρρυθμίσει, δηλαδή είμαστε σε θέση να εξηγιάνουμε τον προπολογισμό μα, τότε δεν έχει καλό μέλλον οτι θελετε αλλα εαν δεν υπαρχει βουλη στην ευρωπη για εσωτερικε μεταρρυθμισει δηλαδη ειμαστε σε θεση να εξηγειάνουμε τον προπολογισμο μα τοτε δεν εχει καλο μελλον η ηπειρο μα και η Λετωνία είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώ τα κάνει σωστά αυτά τα πράγματα κανεί. Δεύτερον, η συζήτηση για τη δημοκρατία που έχουμε. Τι μάθαμε την Κυριακή. 61% των ε, Ελλήνων είναι κατά περαιτέρω περικοπών. Μα είναι τόσο περίεργο αυτό. Αν ψηφίζαμε στη Φιλανδία ένα δημοψήφισμα, τότε εκεί θα μπορεί να έλεγαν οι Φιλανδοί δεν είμαστε διαδεθμένοι να πληρώνουμε τους φόρους μας για τη διάσωση άλλων χωρών της Ελλάδας. Αυτό τι είναι, είναι κακή δημοκρατία, αυτό δεν θέλουν να δώσουν φορολογούμενοι. Τι μάθαμε, ότι υπάρχουν εθνικές προοπτικές, αλλά δεν προωθούν την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι ως ιδέα το ότι καθόμαστε όλοι γύρω γύρω από ένα τραπέζι για να επιτύχουμε συμβασμό. Όχι προκλήσεις, όχι αντιπαράθεση. Συμβασμοί. Γι' αυτό η Κυριακή δεν ήταν καλή ημέρα για την Ευρώπη. Υπέστη βλάβη η Ευρώπη την προηγούμενη Κυριακή. Και οι επιφημίες που ακούσαμε από, την, ε, από διάφορες ακραίες πλευρές για το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι καλές για την Ευρώπη. Κοιτάξτε. Ορισμένοι λένε ότι είναι άδικη η συμφωνία που προτείνεται. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί όλα αυτά τα ε, απογεύματα που προσπάθησε να διαπραγματευτεί με τον ε, Τσίπρα και την ελληνική κυβέρνηση ήταν για να επιτευχθεί μια καλή συμφωνία. Δεν, προ, δεν, προ, δεν προτινόταν περαιτέρω περικοπέ στι συντάξει. Πρότειναν περικοπέ στι στρατιωτικέ δαπάνε και προβλέπονταν 35 δι για την ανάπτυξη Ελλάδα. Και αυτά η ελληνική κυβέρνηση με ευκολία τα απέρριψε. Βεβαίως ήταν μια δίκαιη συμφωνία αυτή που προτινόταν και για μας, αυτή τη στιγμή για την ομάδα μας τουλάχιστον, δεν έχουμε καμία δυνατότητα να δούμε πώ είναι δυνατόν. Δεν έχουμε καμία δυνατότητα να φανταστούμε πόσο παραπέρα θα μπορούσαν να πάνε αυτές οι προτάσεις. Το παιχνίδι του ΣΥΡΙΖΑ είναι υψηλού κινδύνου. Η Ελλάδα ήταν σε μια δύσκολη κατάσταση, η Ελλάδα έκανε πολλές περικοπές, Μειώθηκε ε, το ΑΕΠ, αυτό ήταν σίγουρα μεγάλο βάρος για τη χώρα, αλλά δυστυχώς τους τελευταίους πέντε μήνες προχώρησε ακόμη πολύ περισσότερο η κατάσταση. Υπάρχει έλλειψη φαρμάκων, έχουν κλείσει τράπεζες, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση της Ελλάδας. Και αυτό είναι και ευθύνη του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, αγαπητοί συνάδελφοι. Εάν κοιτάξουμε σήμερα την Ελλάδα, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει διχόνοια σε αυτή τη χώρα. Και αυτό είναι αποτέλεσμα τη κυβερνητική πολιτική του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι καλό απολογισμό αυτό για την Ελλάδα. Και τέλο, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να πω. Η Ευρώπη, και το ξέρουμε όλοι, βασίζεται επί αρχών αλλά και επί κανόνων. Και οι δύο πλευρέ είναι σημαντικέ. Οι αξίε είναι δημοκρατία, αλληλεγγύη και νομίζω ότι η Ευρώπη είναι υπόδειγμα για όλο τον πλανήτη. Από την άλλη μεριά όμω, Ευρώπη σημαίνει και κανόνε και τήρηση των κανόνων. Τήρηση των συμφωνιών, των συμβάσεων που έχουν αποφασιστεί. Και αυτό είναι Ευρώπη και ελπίζω τα επόμενα χρόνια να επανέλθουμε και στην τήρηση αυτής της αρχής. Ότι πρέπει να γίνονται σεβαστοί οι κανόνες. Για την ομάδα των ε, ε, σοσιαλιστών, ο κ. Πιτέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προς τη Λετωνική Προεδρία να πω ότι κινηθήκατε με καλές προθέσεις και με ε, απόλυτη ικανότητα και πετύχατε σημαντικά αποτελέσματα. Σκέφτομαι ιδιαίτερα στην έγκριση του προγράμματος επενδύσεων και των μέτρων για την περιαγωγή. Όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το αίσθημα ανησυχίας που αγγίζει πολλούς από τους πολίτες. Πολλές σύνοδοι κορυφής ε, στην Ευρώπη κατέληξαν σε αποτελέσματα μερικά αποσπασματικά για τη μετανάστευση. Παρουσίασε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά το Συμβούλιο προσπάθησε να το υποβαθμίσει. Τα κράτη-μέλη και όλοι εμείς προσπαθούμε, πρέπει να αναλάβουμε πλήρως τις ευθύνε μας. Και περισσότερο από ποτέ πρέπει να πούμε ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική καμπή. Νομίζω και εγώ ότι δεν υπάρχει εναλλακτική στη συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των πιστωτών της. Δεν μπορώ καν να σκεφτώ το σενάριο έλλειψης συμφωνίας. Διότι αν δεν υπάρξει συνεννόηση, αυτό θα πει ότι ανοίγουμε την πόρτα σε, μια, ε, σε ένα σενάριο, μια περίπτωση καταστροφική που θα θίξει όχι μόνο την σταθερότητα της Ευρωζώνης, αλλά και το μέλλον της Ευρώπης. Συμμερίζομαι λοιπόν πλήρως τη θέση του Πρόεδρου Γιούγκερ. Τον ευχαριστώ για την υποδομητική ε, του αφοσίωση στο να βρεθεί λύση και πρέπει να αξιοποιήσουμε κάθε δευτερόλεπτο μέχρι τέλου για να βρούμε μια συμφωνία με του πιστωτέ. Το αποτέλεσμα τη ελληνική ψήφου για μένα, για όλου μα του Ευρωπαίου ε, τη Δημοκρατία Είναι σαφέ. οι Έλληνε δεν θέλουν να βγουν από το ευρώ. Θέλουν να ε, διαπραγματευτούν μια συμφωνία που να επιτρέπει να οικοδομηθεί ένα μέλλον θετική αξιοπρέπεια. Όλε οι κυβερνήσει τη Ευρωζώνης θα πρέπει να ακούσουν με προσοχή αυτό το μήνυμα και να κάνουν μια προσπάθεια για να ξεπεράσουν την αδιαλαξία, γιατί είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα ο Υπουργό Οικονομικών που χθε είπε ότι το Brexit είναι η μόνη δυνατότητα, του απαντώ προσοχή. Προσοχή, διότι θα αντιταχθούμε σε όποιον ε, θέσει τέτοια τελεσίγραφα και σε όποιον παίζει με το μέλλον της ε, Ευρώπης. Στον Τσίπρα και την κυβέρνησή του θα έπρεπε να πω ότι σήμερα στη Σύνοδο θα πρέπει να έχουμε λογικές προτάσεις. Τώρα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους όλοι. Και είναι απαράδεκτες οι κατηγορίες ενός πρώην Έλληνα Υπουργού προς τους πιστωτές που τους χαρακτήρισε δημοκράτες. Ε, αυτό είναι εύγλωτο. Όλα τα ελληνικά κόμματα έχουν υπογράψει ένα κείμενο συνεννόησης για να καταλήξουμε σε κάτι λογικό. Με μια επικοδομητική προσέγγιση λοιπόν η Σύνοδος απόψε το βράδυ μπορεί να ανοίξει την ε, πόρτα σε μια γέφυρα, ε, ένα πέρασμα που να επιτρέψει οι Έλληνες πολίτες να ανασάνουν και να ε, αξιοποιηθεί και το Ταμείο Διάσωσης θα πρέπει να πάψει αυτός ο τραπεζικός πανικός. Το ελληνικό πιστοτικό σύστημα θα πρέπει να έχει τέτοιες δυνατότητες που να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί. Όπως σωστά είπε ο πρόεδρος ε, Γιούνκερ, ε, κύριε Σούλτς, κύριε Γιούνκερ, για πρόεδρε του Συμβουλίου, αυτή τη στιγμή σε αυτές τις αντικσότητες θέλω να θυμίσω όλους, σε όλους μας ότι μια έξοδος ε, από την, ε, από την ζώνη ευρώ για την Ελλάδα θα ήταν ε, μια πορεία χωρίς επιστροφή. Μπορεί να οδηγηθούμε σε διάλυση, θα πληγεί η υπερηφάνεια όλων μας εάν δεν σώσουμε την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ομάδα ECA ο κύριος Ρόμπερτ Ζήλε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, κυρία Προεδρεύουσα, πρώτα απ' όλα εξ ονόματος της ομάδας να ευχαριστήσω την Προεδρεύουσα του Συμβουλή για την πολύ καλή δουλειά. Πήρε ο κύριος Βέμπερ ε, ε, τα λόγια από το στόμα μου και εγώ ήθελα να επισημάνω την παρουσία γυναικών στις τρεις πρώτες σειρές εδράνων. Δεν υπάρχει ανισότητα μεταξύ των δύο φίλων. Γι' αυτό και τόσο καλό είναι το αποτέλεσμα και τα επιτέμματα αυτής της λειτουργικής Προεδρίας είναι αξιοσημείωτα. Οι συνάδελφοί μου είπαν πολύ καλά λόγια για τα πολιτισμικά προγραμματά και για τα τεχνικά ζητήματα. Η χώρα μου είναι ένας ε, σημαντικός πυλώνας της ε, ε, ποικιλομορφίας της Ευρώπης. Έχουμε επίσης επιτύχει σημαντικά και στον τομέα της ενίας αγοράς. Είχαμε και το πακέτο τηλεπικοινωνιών που θα προωθήσει το ψηφιακό θεματολόγιο. Έχουμε τα ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στα οποία επίση σημειώθηκε πρόοδο και το πακέτο για τις οδικές μεταφορές και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι σημαντικά επιτεύγματα και οδηγούν σε μια νέα πορεία, σε μια νέα κατεύθυνση την Ευρώπη. Έχουμε επίση το EFSE e που το αφήνω λίγο κατά μέρο, δηλαδή το πρόγραμμα επενδύσεων, γιατί κατά την άποψή μου ο ε, κύριος ε, Γιούνκερ έκανε κάποιες ε, ε προτάσει, κάποιε υποσχέσει για ένα εξάμεινο, αλλά αυτά σίγουρα δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσα σε έξι μήνες. Έχουμε νέες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν θα ήθελα να βιώσω ότι ενώ έχουμε αυτό το θέμα της γεωγραφικής ουδετερότητας, τελικά να μιλάμε για γεωγραφική συγκέντρωση η πραγματική προτεραιότητα όμως λιτωνικής προεδρίας και ένα σταθμό, θα έλεγα, ήταν η Σύνοδος Κορυφής Εταιρικής ε, Σχέσης προς Ανατολάς. Έχουμε τους Ουκρανούς, τους Γεωργιανούς, που στράφηκαν προς, το, προς τη Δύση για το μέλλον τους ε, και ήταν ε, ε, ίσως και κάπως, πήραν και κάποιο ρίσκο κάνοντας αυτό. Νιώθουν απογοητευμένοι ενδεχομένως. Οι Ευρωπαίοι δεν θέλησαν να προχωρήσουν σε μια πιο καταμέτωπο σύγκριση με τη Ρωσία. Πιστεύω ότι διαφορετικές προτεραιότητες ε, θα έπρεπε να είχαμε ε, υποστηρίξει και σε ό,τι αφορά τώρα το ελληνικό ζήτημα. Συμφωνώ ότι το θέμα είναι πάρα πολύ ε, πολύπλοκο. Δεν είναι απλό. Το είπε και ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί ε, στη Λετωνία περάσαμε ένα πρόγραμμα λιτότητα και γι' αυτό θέλουμε και για την Ελλάδα μια δίκαιη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσίλε. Από πλευρά ο κύριο Φερχόφσταντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω όσα είπατε είναι απολύτως αληθή, κύριε Γιούγκερ. Ας επανέλθουμε ε, στην ε, κοινή λογική διότι τις τελευταίες δύο-τρεις μέρες άκουσα κάποιες φωνές λογικής για την ελληνική κρίση, αλλά κάποιοι άλλοι μιλάνε για τον Brexit σαν να μην πρόκειται για πρόβλημα. Δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα όμως, μιλάμε για τη δυνατότητα να έχουμε υγιή νομισματική ένωση, να είμαστε ικανοί ως νομισματική ένωση να λύσουμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Μιλάμε για για ένα ιστορικό ε, χρέος 300 δις. Εδώ ε, μιλάμε για, ένα, ε, για μια ε, νομισματική ένωση με 303 με 15-3 ΑΕΠ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, να μην μπορούμε να λύσουμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ, ας επανέλθουμε στην κοινή λογική και να μην λέμε ότι να είναι το ίδιο και για το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Πρώτα απ' όλα προτείνεται μια συμφωνία ε, στον Τραπέζι των μετά δημοσιεύουν ένα κείμενο που λένε ότι η συμφωνία αυτή δεν είναι βιώσιμη. Τι επιθυμότητα είναι αυτή. Και νομίζω, κύριε Γιούνκερ, πρέπει να βρούμε μια νέα προσέγγιση. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν πετυχαίνει η λύση που έχουμε προτείνει ως τώρα για την ελληνική κρίση. Και αυτό ε, το βλέπω εγώ, ε, ισχύει και για μένα και ισχύει για όλες τις πολιτικές ελίτ στην Ευρώπη. Ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει σαφώς να προτείνει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Όχι μόνο μέτρα λογιστικής όπως τώρα έχουμε στο τραπέζι ε, των διαπραγματεύσεων, μια πραγματική μεταρρύθμιση, ένα του χρέου. Πρέπει να πάψει το σύστημα που ισχύει ω τώρα. Δεν είναι βιώσιμο σήμερα. Πρέπει να πάψει η διαφθορά στη χώρα. Να μειωθεί ο δημόσιο τομέα, ο οποίο είναι τεράστιο, με 800.000 ε, δημόσιου υπαλλήλου αυτή τη στιγμή. Κάτι πρέπει να προταθεί. Ε, να σωθούν οι δημόσιε τράπεζε με ένα νομό ιδιωτικό τομέα. Και για τι αγορέ. Πρέπει να βγει η χώρα στι αγορέ. Αυτό πρέπει να κάνει τώρα. Να μα πει τι είναι οι προτάσει του. Ξέφυγε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Α προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το χρέο στην Ευρώπη όμω από κοινού. Εάν είχαμε δημιουργήσει ένα ταμείο διάσωση ε, πριν από λίγα χρόνια, δεν, είχαμε, δεν θα είχαμε ε, τα σημερινά προβλήματα. Θα είχαμε ένα πραγματικό εργαλείο για να λύσουμε και να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Α είμαστε λοιπόν έτοιμοι, διότι δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Εάν δεν ε, ε, βοηθήσουμε του Έλληνε, αν δεν βοηθήσουμε την ελληνική κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τα κατεπήγοντα μέτρα που έχουν προβλεφθεί και αν δεν βοηθήσουμε απευθεία του Έλληνες πολίτε και τις ελληνικέ οικογένειε ε, τι ερχόμενε εβδομάδε και μήνες, τι θα κάνουμε. Ε, καλή τύχη για απόψε. Ε, Ευχαριστώ για την ομάδα των Πρασίνων η κυρία Χάμς. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου κυρίε και κύριοι, όντως, όντως ισχύει και πραγματικά με αγωνία περιμένω να δω τι θα πει ο κύριος Σύπρα σήμερα για την Ελλάδα. Αλλά είναι μεγάλη πρόκληση και το όχι να εκπροσωπήσει κανείς και το ναι. Γιατί το πρώτο του καθήκον είναι η χώρα του να είναι και πάλι ενωμένη γιατί μόνο μια ενωμένη Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί επιτυχώς στις Βρυξέλλες. Οι εκκλήσεις προς τον κύριο Τσίπρα που έγιναν τις τελευταίες μέρες πολλές τις ημερίζομαι αλλά σήμερα πρέπει επίσης να πω ότι υπάρχουν και ορισμένες ε, εκκλήσεις προς την κυρία Μέρκελ την οποία, τις οποίες δεν δέχομαι και είναι καλός ο τόνος της κυρίας Γιούνκερ. Η Bild σήμερα λέει ότι αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι μια σιδηρά καγκελάριος. Μα είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Θα ήθελα και οι Γερμανοί να θυμηθούν ότι εμείς όταν ε, αν είχαμε πάντα ενώπιόν μας σιδηρούς γείτονες δεν θα είχαμε αυτή τη Γερμανία, δεν θα είχαμε αυτά τα ευρωπαϊκά έθνη γιατί η Γερμανία έχει μια πολύ συγκεκριμένη ευθύνη. Κύριε Γιούγκερ, νομίζω ότι και τα δύο είναι σαφή. Από τη μία πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις οι οποίες αναφέρονται και στο κείμενο του Δουνουτού. Δεν μιλάει το κείμενο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη μη βιωσιμότητα του χρέους. Το κείμενο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κάνει σαφείς εκκλήσεις για τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην Ελλάδα. Από την άλλη μεριά πρέπει να γίνει βιώσιμο το χρέος της Ελλάδας. Και κυρία Πρόεδρε, η χώρα, η χώρα σας με ενθουσίασε, γιατί η χώρα σας είναι ακόμη σε ανάπτυξη και έχει πολλά προβλήματα, αλλά με ιδιαίτερα φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση. Θα ήθελα λοιπόν αυτοί οι νέοι Λετωνοί, οι νέοι από τις χώρες Βαλτικής και οι νέοι Έλληνες να μπορέσουν να συνοηθούν για το τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία αντί να αντιπαρατίθενται. Πιστεύω μάλιστα ότι οι νέες, κυρίως μικρές χώρες, μπορούν να παίξουν ένα ρόλο γέφυρα σε όλη αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ για την Προεδρία σας και σας εύχομαι και σας και στη χώρα σας και στην Ευρώπη καλή τύχη και επιτυχία. Ευχαριστώ για την ομάδα EFTD, ο κύριος Νάτορος. Κύριε κύριε Πρωθυπουργέ, είπατε ότι η Λεπτονική Προεδρία ε, έκανε καλά τη δουλειά της. Μα τι ακούω εδώ πέρα. Γκίλτ the lily που λέμε στην Αγγλία. Χρυσώνουμε το χάπι εδώ, δεν θα πρέπει αντί να οριοποιούμε την κατάσταση να λέμε την αλήθεια. Η Προεδρία σας ήταν μια καταστροφή ανευπροηγουμένου. Δεν μπορεί να μετριαστεί αυτή η καταστροφή. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, για να δούμε τι συμβαίνει, συνεχίζει να γίνεται τη Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Ε, ε, χορεύει γύρω-γύρω στην Ουκρανία και κανεί δεν κάνει τίποτα. Έχουμε 500.000 μετανάστε στη Μεσόγειο και άλλοι 500.000 που περιμένουν. Και η Eurojust χθες παραδέχθηκε ότι το ίσις στέλνει ε, τζιχαντιστές στην Ήπειρό μας και απ' την άλλη έχουμε την Ελλάδα που ενδεχομένως να εγκαταλείψει το ευρώ. Και όλα αυτά ε, υπό το δικό σας βλέμμα έγιναν, ε, κύρια Πρωθυπουργέ. Δεν είναι και τόσο καλό αυτό το αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν κάνατε ουσιαστικά τίποτα ε, απλά σιγοτραγουδούσατε βλέποντας όλα αυτά να συμβαίνουν και ως ευρωσκεπτικιστής ε, εγώ θα ήθελα ε, η Λετωνία να παραμείνει στην Προεδρία για έξι μήνες ακόμη γιατί έτσι θα καταρρεύσει σε έξι μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση εντελώς. Και τώρα για το κόμμα ΕΝΕΦ, e Ευρώπη των Εθνών και της ε, Ελευθερίας, ο κ. Μπονάνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στρέφομαι στην Υπουργό, την Προεδρία που μόλις τελειώνει Συγχαρητήρια. Αλλά επειδή είχαμε τρει γυναίκε, δεν πάνε όλα καλά. Υπάρχουν ε, γυναίκε που πάνε καλά ε, και λιγότερο. Το ίδιο και για του άνδρε. Δεν σημαίνει ότι τρει γυναίκε είναι καλύτερε από τρει άνδρε. Α αφήσουμε λοιπόν την υποκρισία κατά μέρο. Σε ό,τι αφορά τώρα τον ε, κύριο Γιούνκερ, τον βλέπω εδώ πρώτη φορά από αυτή τη θέση και θέλω να του κάνω τι εξή ερωτήσεις. Έχετε πάει να αγοράσετε ένα λίτρο γάλα, ένα κιλό ψωμί και ένα λίτρο βενζίνη. Τι γίνεται με τα χρήματα που πάνε στις πολυεθνικές, στις μεγάλες τράπεζες και μένουν στις τσέπες των ίδιων. Ο λαός, ο κόσμος δεν νοιάζεται για αυτά. Χρειάζεται άλλες απαντήσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή είναι η σημαία της Γερμανίας και αυτή της Ευρώπης. Δεν θέλω να πεθάνω ως Γερμανός ή Ευρώπη ή Γερμανία. Ιδάλω, εάν συνεχίσουμε έτσι, η Ευρώπη μικραίνει. Μικραίνει όμω και για τη Γερμανία. Η Γερμανία είναι αυτή που πρέπει να, ε, να μικρύνει. Δεν μπορεί να διατάζει όλη την Ευρώπη. Ε, έχουμε ήδη δει τι έφερε στην Ευρώπη ο ναζισμό. Δεν θέλουμε τώρα λοιπόν οικονομικό ναζισμό. Θα πρέπει, ναζισμό. Θα πρέπει να αλλάξουμε λιγάκι την πορεία των πραγμάτων. Ιδάλω, κύριε Γιούνκερ, 100 δι επενδύσει. Πού θα πάνε. Βλέπετε εδώ άλλες, άλλες, άλλα παραδείγματα. Το χαρτί υγείας από τη μια και το ευρώ από την άλλη. Έχουν καταντήσει να είναι το ίδιο με τη δουλειά σας. Δεν πάει πουθενά η Ευρώπη. Δεν κάνετε αυτό που ενδιαφέρει το λαό. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να παρετηθείτε. Να παρετηθείτε και να ζητήσετε συγγνώμη από την Ελλάδα για όσα κάνετε. Να ζητήσετε συγγνώμη από όλη την Ευρώπη. Διότι με τις οικονομικές σας επιταγές μας οδηγείτε σε ε, σύγκρουση, σε ε, αυτοκτονίες, σε λάθρο άλλο θέλετε. Ευχαριστώ κύριε Μπονάνο. Και τώρα... Και τώρα... Η κυρία Μόρβαη, μία εγγεγραμμένη. Ευχαριστώ πολύ. Η προέρχομαι από ένα έθνος το οποίο αντιμετωπίζεται ως δευτέρας κατηγορίας και γι' αυτό Περίμενα με πολλή ε, προσδοκία και παρακολούθησα με πολύ ενδιαφέρον την Λετωνική Προεδρία. Και με βάση τη σημερινή συζήτηση μπορώ να πω ότι εκπρόσωπος ε, του Συμβουλίου ε, είχε τον ίδιο τόνο, την ίδια επιχειρηματολογία, όπως και ο κύριος Γιούγκερ. Ευτυχώς κανείς δεν επιχείρησε να δείρει κανέναν άλλο εδώ μέσα σήμερα. ο κύριος Γιούγκερ, ο οποίος είναι από το Λουξεμβούργο, και οι άλλοι πολιτικοί της ε, ε, Δυτικής Ευρώπης, αυτοί που είναι ε, από τις χώρες της πρώτης σειράς, που είναι ε, από ευημερούσες χώρες, μιλάνε με ήρεμο τρόπο, γιατί δεν έχουν ιδέα για τα προβλήματα που υφίστανται οι άνθρωποι είπαν ότι θα μας μιλήσουν για την κατάσταση ανάγκης και τα προβλήματα που έχει η, η Ελλάδα, οι πρώην κομμουνιστικές χώρες, αλλά δεν έχουν ιδέα για όλα αυτά τα θέματα. Δεν έχουν καμία προσωπική εμπειρία. Δεν καταλαβαίνουν γιατί πολλοί χρειάζεται να καταλήψουν τη χώρα τους, ακόμη και από τις δικές τους τις χώρες, ακόμη και από τη δική μου χώρα, αλλά βέβαια κυρίως από την Ελλάδα ή από άλλες χώρες του Νότου. Περί τίνος πρόκειται. Πόσο θα κρατήσει ακόμη αυτή η διάκριση, η μεταξύ πρώτης και δεύτερης κατηγορίας ε, κρατών. Αυτό έπρεπε να έχει πει η Λετωνική Προεδρία. Αυτό περιμένουν οι πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, για άλλη μια φορά, ο κύριος Γιούγκερ, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, Κυρίε και κύριοι, να πω στο τέλο αυτής της συζήτηση ότι αυτοί οι οποίοι χωρί λόγο προσβάλλουν τη Λετωνική Προεδρία ασφάλουν διότι ήταν εξαιρετική η δουλειά της Λετωνικής Προεδρίας. Γι' αυτό και αντιπαρατήθαμε σε αυτές τις αβάσιμες, άδικες και αδικαιολόγητες κατηγορίες και επικρίσεις. Και για να επανέλθω στο ζήτημα που μας απασχολεί σήμερα, ή την Ελλάδα, θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη βούληση να κάνει πάνω το δυνατό για την επίτευξη συμφωνίας. Και να πω ότι η Ευρώπη δεν αποτελείται από μία μόνο δημοκρατία, αλλά από 19 δημοκρατίε και θα πρέπει σίγουρα να προσπίσουμε τα συμφέροντα τη Ευρωζώνη στο σύνολό τη. Καθώ επίση και να σεβαστούμε ε, και τις επιλογές ε, και τη βούληση και των 18 άλλων δημοκρατιών. Γιατί μια δημοκρατία δεν αξίζει περισσότερο από τις άλλες δημοκρατίες. Ένας πολίτης ε, είναι παντού το ίδιο. Ένας πολίτης. Σταματήστε επίσης τη φλιαρία αυτή που μου ε, λέτε συνεχώς ότι κοιτάζω το τηλέφωνό μου διότι έχω ε, ανταλλαγή μηνυμάτων με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, texting όπως το λέμε στα γαλλοαγγλικά. Δεν ξέρω αν εσείς ε, έχετε δυνατόν να το κάνετε. Κάνω τη δουλειά μου, σταματήστε λοιπόν να φλιαρείτε ανοήτως. Επίσης, το να δίνουμε την ε, ιδέα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για για ε, την Ευρώπη ότι είμαστε εδώ σε μια λέσχη ε, χρυσή και ότι δεν βλέπουμε πώς ζουν πραγματικά οι πολίτες, ότι είμαστε σε ένα ξελεφάντινο πύργο. Αυτό είναι στοιχειώδης λαϊκισμός, είναι μια ανθυγιεινή πρακτική και ρητορική. Εγώ κάθε εβδομάδα έχω επαφές με τους Έλληνες πολίτες και δεν μιλώ μόνο για την κυβέρνηση ή τα άλλα πολιτικά πολιτικά κόμματα, μιλώ για Έλληνες πολίτε με τους οποίους έχω επαφές και πρέπει να σας πω ότι είμαι μεταξύ αυτών που ασχολήθηκαν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο με τις συνθήκε διαβίωση και εργασίας των Ελλήνων πολιτών. Μην δίνετε λοιπόν την εντύπωση ότι είμαστε μακριά από τους Έλληνες πολίτες ή από τους άλλου πολίτε και για να ασχοληθώ ακριβώς ε, με την καθημερινή πραγματικότητα των Ελλήνων πολιτών να σας πω ότι δεν ξεχνώ και την καθημερινότητα των άλλων χωρών. Ανεργία υπάρχει παντού στην Ευρώπη, φτώχεια υπάρχει παντού στην Ευρώπη. Η κατώτατη ε, κοινωνική ε, μισθή και η κατώτατη ελάχιστη μισθή είναι σε κάποιες χώρες μικρότερη από το κατώτατο μισθό στην Ελλάδα. Υπάρχουν ε, επίσης συνθήκες διαβίωσης σε χώρες που είναι χειρότερες ε, από ό,τι στην Ελλάδα. Πρέπει να βλέπουμε λοιπόν συνολικά την πραγματικότητα ε, και να μην πέφτουμε στην παγίδα της δημαγωγίας και του λαϊκισμού. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πραγματικά πολλοί εξ αυτών ε, ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και άλλους πολίτες, γιατί είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε και την Ελλάδα και την Ευρώπη. Να μην ξεχνάμε την Ελλάδα, αλλά να μην ξεχνάμε και την υπόλοιπη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Κύριε Γιούγκα. Κύριε εκεί. Κύριε Δημάζη, να βάλετε σωστά ε, αυτό το χαρτί που έχετε, γιατί εγώ καταλαβαίνω ίζο από αυτό που βλέπω να έχετε βάλει εκεί. Κυρίες και κύριοι, πριν δώσω το λόγο στην κυρία Στραουγιούμα, Κυρία Στραουγιούμα, πριν σας δώσω και πάλι το λόγο, θα ήθελα, νομίζω από πλευρά τη μεγάλη πλειοψηφία των μελών του σώματο, ότι σα ευχαριστούμε πάρα πολύ και προσωπικά για την ε, θαυμάσια προσπάθεια που κάνατε, για την ε, πολύ σκληρή εργασία που επιτελέσατε. Νομίζω ότι ε, για μια μικρή χώρα είναι πολύ μεγάλη η πρόκληση να ηγηθούν τη Προεδρία του Συμβουλίου. Ο τρόπο με, τον οποίο, με τον οποίο επιτελέσατε κάθε κοντά σα ήταν υποδειγματικό και γι' αυτό σα ευχαριστώ πολύ. Η κυρία λοιπόν. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ήταν μεγάλη μου χαρά να μπορούμε να συζητήσουμε τα επιτεύγματα της Λετωνικής Προεδρίας. Γνωρίζω ωστόσο ότι το βασικό θέμα σήμερα είναι η Ελλάδα. Έχει καταλάβει τις σκέψεις και το νου όλων μας Αναμφίβολα η κατάσταση στην Ελλάδα είναι ε, πρώτη προτεραιότητα στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε στηρίξει κάθε προσπάθεια για να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα στις συνομιλίες Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδας. Εντός ολίγου θα συναντηθούν οι Υπουργοί Οικονομικών και εγώ ίδια θα ταξιδέψω απευθείας από το Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχω στην έκτακτη σύνοδο κορυφής. Και όπως είπε και ο Ζαν Κλοντ, περιμένουμε οι συγκεκριμένες προτάσεις από την Ελλάδα με ένα όραμα, μία άποψη για το πώς η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να συμβαδίσουν. Είναι σημαντικό να επικεντρώνεται κανείς στο πώς να τακτοποιεί ε, ε, το δικό του ε, σπίτι, αλλά και να μην χάνεται χρόνος. Το επαναλαμβάνω, χρόνος είναι πολύτιμος. Κάθε μέρα που περνάει είναι μία απώλεια. Ελπίζω λοιπόν ότι ο νέος Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας και ο Πρωθυπουργός της θα φέρουν στο τραπέζι των δημοτεύσεων επικοδομητικές προτάσεις. Και εν είδη συμπεράσματος να ευχαριστήσω ξανά το Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι μαζί μπορέσαμε να βρούμε λύσεις στις σημαντικότατες προκλήσεις που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ελπίζω ότι το τελευταίο εξάμεινο γνωρίσατε μια μικρή χώρα στο βορρά της Ευρώπης, τον πολιτισμό μας, τις παραδόσεις μας, τις δυνατότητές μας. Σας ευχαριστώ και θα σας δούμε και πάλι στην επόμενη Προεδρία της Λετωνίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στραβιούμε. Ε, ο κύριος Χλέζος με παρακάλεσε να του δώσω το λόγο γιατί σήμερα είναι η τελευταία μέρα που συμμετέχει στην Ολομέλεια. Νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο μπορώ γι να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γλέζο για μια προσωπική δήλωση. Πρώτον μεν ήρξω του λόγου ψευδός ξένε ζητών τύραννων ενθάδε ενθάδε ούγαρ άρχεται ενός προσανδρός αλελευθέρα πόλης. Δήμος δανάσι διαδοχέσιν εν μέρη ενιαυσίασιν. Οχι το πλούτο διδός το πλήστον, αλλά χοπένης έχων ίσον. Είναι λόγια του Θησέα όταν ο Θηβαίος ζήτησε ποιος είναι τύρανος στην Αθήνα και επέλεξα αυτό το σημείο από τα αρχαία ελληνικά και θα επιλέξω κι άλλο ένα σημείο από τα λατινικά που πιστεύω το γνωρίζει πολύ καλά ο πρόεδρος μας ο Μάρτιν Σούλτς. Ο Θωμάς ο Κουινάτος είπε «Τίμεο χόμινεμ ουνίους λίμπρι» και και τα δύο αυτά κείμενα είναι η απάντησή μου και για την λετονική θητεία και για όλο το κοινοβούλιο και για σας προσωπικά αγαπητέ πρόεδρε. ευχαριστώ. Το επόμενο θέμα της μέρες διάταξης